στη Σομαλία και περνάμε στις παρεμβάσεις των συντακτών ο κύριος Κοράο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σομαλία εξακολουθεί να γνωρίζει πολλού πολλούς θανάτους και εκτοπισμούς άοπλων. Ε, τον Ιούλιο η πατιαρμοστία το ΙΕ ανέφερε ότι ε, καταναγκαστικές εκδιώξεις λόγω των συνεχιζόμενων σειράξεων ε, οδήγησε σε εκτοπισμούς 28.000 ανθρώπων. Διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν σοβαρές καταχρήσεις κατά των ανθρώπων που ζουν σε επίσημους καταβλισμούς εκτοπισμένων και σε κυβερνητικές περιοχές συμπεριλαμβανομένου βιασμού και αναγκαστικών ε, ε, εκδιώξεων ή εξώσεων Επίσης οι δημοσιογράφοι απειλούνται, ε, κρατούνται παράνομα και δεν ε, τους ε, παρέχεται καμία εγγύηση δίκαιης δίκης. Αυτό είναι πολύ σοβαρή ανησυχία, ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος ότι θα γίνουν εκλογές κανονικά σύντομα. Πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια για την προστασία του πληθυσμού, όπως θα πρέπει και να βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Σομαλίας στην εργασία της για δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουμε υπόψη την κατάσταση και να την παρακολουθούμε ώστε να ε, μην γίνονται παραβιάσεις. Ελπίζουμε πως αυτό το κοινό ψήφισμα θα βοηθήσει σε αυτό. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, πέντε χρόνια μετά ε, την, την εκδίωξη της Αλσαμπάφ στο Μογκαντήσου έχει βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας. Ε, οδεύουμε προς δημοκρατικές εκλογές. Αυτές οι εξελίξεις σίγουρα είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, η εικόνα είναι ανάμεικτη ακόμη. Χθε οι ηγέτες των γειτονικών χωρών πήγαν σε μια διάσκεψη κορυφή στο Μογκαντήσου για πρώτη φορά <clears throat> μέσα σε δεκαετίες. Αυτό όμως δεν μας κάνει να παραγνωρίζουμε το γεγονό ότι πριν από δύο εβδομάδε. τουλάχιστον δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια τρομοκρατική η επίθεση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Πρέπει να δώσουμε ε, περαιτέρω ενίσχυση στην Άμυσο. Αυτό είναι απαραίτητο, είναι ζωτικό. Αλλά <clears throat> και τις προσπάθειες ε, της ε, αποστολής για την καταπολέμηση της πειρατείας στις <clears throat> ακτές της Σομαλίας από την ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο τη πολιτική ΚΕΠΑ. Επίση, τι γίνεται στη Σομαλιλάνδη ε, και πώ συνεργάζεται με την κυβέρνηση της, ε, του Μογκαντήσου. Υπάρχει μια ένωση, η οποία όμω με, με δημοψήφισμα δεν έχει επικυρωθεί. Για μια ελεύθερη Σομαλιλάνδη προηγούνται οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να προηγηθούν συνομιλίες δημοκρατικές. Στο κέρα Αφρική πρέπει να επικρατήσει χρόνια ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ κύριο Σκέλαμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι στρατηγική θέση της Σομαλίας. Η σταθερότητα, η προστασία από τρομοκρατικές επιθέσεις είναι ζωτική σημασίας. Μετά από δύο δεκαετίες ε, εμφύλου πολέμου και την τρομοκρατία που ασκεί ο οργάνος Βελτίωση έχουμε, αλλά δεν έχουμε καμιά εγγύηση 16 Ιουλίου και Αύγουστο επίση 24 έγιναν δύο τρομοκρατικέ εκθέσει που δείχνουν ότι η Al-Shabaab ε, ακόμη ε, είναι ενεργή. Ε, πρέπει αυτά τα οποία ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια να συνεχιστούν. Έχουμε τι εκλογέ το 2020. Τα πολιτικά κόμματα δημιουργούνται, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ελευθερία έκφρασης και να μπορεί και η ε, Διεθνής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να έχει το ρόλο της. Θα είναι σημαντική και δράση της ειρηνευτικής αποστολής δυστυχώ, Δυστυχώς ακόμη υπάρχει μεγάλη επισφάλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει όμως ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη και τούμπαλιν. Πρέπει να σπάσει ο φαύλο κύκλο και αυτό απαιτεί κοινέ προσπάθειε από την Εθνική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Αράντζοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από δεκαετίε ε, σειράξεων εξακολουθεί να υποφέρει ο λαός Σομαλίας. Ε, πράγματι ε, έχουν κάπως συγκρατηθεί τα προβλήματα από πριν από 10 χρόνια, σε σχέση με τότε έγινε πριν από 10 χρόνια, όμως δεν νιώθουν ασφαλείς Σομαλοί. <clears throat> μόνο με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δυνατότητα, θα έχει την εξουσία να εγγυάται την προστασία και τα δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών και την οποία θα τη συμπληρώνουν ε, νόμιμοι θεσμοί που θα στηρίζουν το κράτος δικαίου. Οι επικείμενες ε, εκλογές θα πρέπει να είναι διαφανείς, θα πρέπει να είναι δίκαιες και είναι ένα πρώτο βήμα προς το στόχο αυτό. Η Σομαλία διέρχεται μια σημαντική πολιτική μετάβαση, έναν μετασχηματισμό και θα πρέπει η εθνική κοινότητα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται. Γιατί αν αποσυρθεί και η ειρηνευτική αποστολή, η πρόοδο ε, αυτή θα τεθεί σε κίνδυνο. Δεν θέλουμε η Σομαλία να πέσει στα χέρια των τρομοκρατών. Ευχαριστώ. Σεμπαστιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι αβίωτη κατάσταση στη Σομαλία. Έχουμε τρομοκρατικέ ομάδε όπω την Al-Shabaab. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Ε, και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπιστέντε ή και πολλού πρόσφυγε σε γειτονικέ χώρε. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τρομοκρατία, ε, λέει η κυβέρνηση. Όμω, τι κάνει, προσάγει ε, δημοσιογράφου, μπλοκάρει την πρόσβαση στο ίντερνετ και το καθεξή. Ε, ούτε και τα δικαστήρια είναι αξιόπιστα για να κρίνουν αυτού που έχουν μπει φυλακή. Ε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Είναι τεράστιο, τεράστια ανθρώπινη τραγωδία με βασικά θέματα τα παιδιά, τα οποία τα στρατολογούν οι διάφορες φράξεις, οι διάφορες ε, ομάδες. Έχουμε το Ταμείο Ανάπτυξης Βοήθειας την Ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κάνει κάτι. Εμείς ζητούμε όμως μεγαλύτερη ε, εμπλοκή και έλεγχο για την αποτελεσματική χρήση αυτών των κονδυλίων. Το ψήφισμα είναι ισορροπημένο γιατί καταγγέλει και τις καταχρήσεις ε, των δυνάμεων που είναι εκεί υποτίθεται για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα όπως είναι η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης Ομαλία. Έχουμε σεξουαλική κακοποίηση, ε, χρησιμοποίηση γυναικών ε, ως όπλο σε αυτή την σύραξη. Επίσης δεν θέλουμε να πέσει στη λύθη η Σομαλία. Είναι μια σημαντική χώρα για τα εξωτερικά θέματα. Πρέπει να παραμείνει και επίσης θα πρέπει να απευθύνουμε σαφή έκκληση στι χώρε που δέχονται τις πρόσφυγες Σομαλία να είναι και συνεπεί και ρεαλιστέ, Να, να, να μην επιβάλλουν αυτού του ανθρώπου να επιστρέψουν στι χώρε που κάθε άλλο παρασφαλή είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Σεμπαστιά, έχετε μία γαλάζια κάρτα. Θα θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ευχαρίστω. Ο κύριος Φρουντζούλικα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε κύριε Σεμπαστιά. Πράγματι είναι ε, πάρα πολύ ε, άσχημη κατάσταση. Στην Σομαλία υπάρχουν δολοφονίες παιδιών πάνω από χίλια παιδιά έχασαν τη ζωή τους πέρυσι. Είναι ο Επίτροπος Τελιανίδης μαζί μας σήμερα. Δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα υπέρ των παιδιών της Σομαλίας πρόγραμμα επαναλαμβάνω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία και την υγεία κυρίω των παιδιών από τη Σομαλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Συμφωνώ μαζί σα και οφείλω να συμφωνήσω μαζί σα γιατί αυτό είναι προτεραιότητα για μα και πρέπει να είναι προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φροντίσει τα παιδιά αυτά που, στρατολογούν, ε, που στρατολογούνται και πολεμούν σε αυτόν τον ε, πόλεμο ω ε, όπλα και οι οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους ε, που δεν μπορούν να μεγαλώσουν ως ε, φυσιολογικοί ενήλικοι σε αυτή τη χώρα. Φυσικά και είναι προτεραιότητα για, το μέλλον, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το μέλλον των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ένοπλη σύραξη που εδώ και χρόνο πλήττει τη Σομαλία συνεχίζει να δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό παρά τις δεσμεύσεις ε, της κυβέρνησης Όνολ, η, της κυβέρνησης Ομαλίας, η κατάσταση οδηγεί, εμποδίζει την, την χώρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Οι δημοσιογράφοι ε, κρατούνται σύμφωνα με κανόνες που δεν είναι σύμφωνοι προ αυτού τη διεθνού των ε, ε, Ιανουάριο του 2006 ο πρόεδρος της Ομαλίας υπογράψε μια νομοθεσία για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης που πέρα απέχει από τα διεθνή πρότυπα. Είναι σωστό να ζητήσουμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε διεθνέ επίπεδο ώστε η κυβέρνηση της Σομαλίας να προστατεύσει τους δημοσιογράφους και έτσι ώστε να υπάρχει ελευθεροτυπία και ελεύθερη ενημέρωση και εν γέννη να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν ε, παραβιαστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι, 38% του πληθυσμού δηλαδή στη Σομαλία ζουν ε, διαρκώς ε, ε, διοκόμενοι ή αναγκαστικά εκδιοκόμενοι και μετακινούμενοι. Και αυτό οφείλεται στην αστάθεια και τη βία όπου πειρατές και τρομοκρατικές ομάδες λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Θα πρέπει όλα αυτά να περιοριστούν. Η στρατιωτική αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης πολλές φορές συνεργάζεται και διονύζει αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να προωθηθούν ε, βέβαια ε, δημόσιες πολιτικές όμως ε, η δική μας στήριξη, η σε στρατιωτικές ομάδες ανταποκρίνεται μόνο σε γεωστρατηγικά συμφέροντα και εμπορικά συμφέροντα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς όπως θυμίζει και το ψήφισμα. Η σταθερότητα και η ειρήνη μπορούν μόνο να επιτευχθούν μέσω της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης και των πολιτικών που βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές όπου η εξωπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, γίνονται απόλυτα σεβαστά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σβόμποτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, εδώ μιλάμε για ένα κράτος που τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαλυθεί, έχει διαπορδιαρθωθεί τελείως και του οποίου οι πολίτες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το σεβασμό ουδήποτε δικαιώματός του Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να εξασφαλιστεί η ελάχιστη τουλάχιστον ασφάλεια, ώστε να μην ε, συνεχίσει άλλο η υπονομεύση των θεμελίων της κοινωνίας και να αρχίσει η ανοικοδόμηση δυνατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να επιτρέψει στην ε, Σομαλία να επιστρέψει σε μια ομαλότητα που θα επιτρέψει το κράτος να επιτελεί τα καθήκοντά του έστω τα ελάχιστα. Όταν υπάρχουν ε, ιδιωτικοί στρατοί που ε, ελέγχουν κάποιες περιοχές και που απειλούν τη ζωή των κατοίκων τους, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να ε, ξαναγυρίσει στη διεθνή κοινότητα και σε μια λειτουργία κράτου στη Σομαλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζίλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουν εκλογέ φέτο στη Σομαλία, άρα διέρχονται μια κρίσιμη περίοδο μετάβαση και είναι απαραίτητο να μην χάσει το ραντεβού με την ιστορία. Η αδίποτε όμως εκλογική αναμέτρηση δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση αν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν δεν εξασφαλίζεται ένας ελάχιστος βαθμός σταθερότητας η σταθερότητα. Οι αποστολές ειρηνευτικές της Αφρικανικής Ένωσης πρέπει να επιτελούν το καθήκον τους, να προστατεύουν δηλαδή τους ε, αμάχους και να ε, μην εκτίθεται σε ουδεμία κατηγορία είτε βιασμών είτε βιοπρικιών εις βάρος αμάχων. Υπάρχουν προγράμματα παρακολούθησης, υπάρχουν έρευνες από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει όλα αυτά να αξιοποιηθούν. Επίσης καλώ τις αρχές της Σομαλίας, περιφερειακές και εθνικές, ε, να εξασφαλίσουν την ε, ε, προστασία των δημοσιογράφων που απειλούνται και πολλές φορές απάγονται φωνεύονται από ακραία στοιχεία όπως την Al-Shabaab. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στα, μέια, στα, στα μέσα Ιουλίου και Αυγούστου η Ελ Σαμπάμπ ήταν υπεύθυνη για πολλές ε, δολοφονικές επιθέσεις στη Σομαλία που, και μάλιστα μια από αυτές ήταν κατά μιας βάσης της Αφρικανικής Ένωσης. Εκεί σκοτώθηκαν και οι υπάλληλοι του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι γίνεται αγώνας κατά της Αλσαμπάμπ και άλλων ομάδων, ενόπλων ομάδων και αυτό βασικά το έχει αναλάβει η Αφρικανική Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν λοιπόν όλα να συνδυαστούν με όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο βασικός χρηματοδότης ε, της ε, Αφρικανικής Ένωσης έχει υποσχεθεί 200 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 και θα πρέπει αυτή η στήριξη να ενισχυθεί αλλά σε αντιστάθμισμα χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηρίζει μάλλον δεν μπορεί να ανέχεται οι ειρηνευτικέ δυνάμεις να επέφτουν θύματα αδιάκριτων ε, επιθέσεων, ε, ε, βίας, σεξουαλικής βίας. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν όλα αυτά τα εγκλήματα και οι ενδεχόμενοι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε μόνο δύο λεπτά για το Catch the Eye για τη Σομαλία, οπότε μπορώ να δώσω μόνο δύο φορές το λόγο. Ο κύριος Πόσπισιλ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου και είμαι ικανοποιημένος που συζητούμε τη Σομαλία σήμερα διότι όπως προείπαν συνάδελφοί μου, περιμένουμε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο Κοινοβούλιο τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έπειτα έχουμε τις εκλογές και πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ιδίω τα παιδιά της ε, Σομαλής που υποφέρουν, να στηρίξουμε και οικονομικά. Σωστό είναι αυτό. Όμως, ως προϋπόθεση θα πρέπει να είναι ε, η χώρα να ακολουθεί στην οδό της δημοκρατίας. Να δούμε τι θα γίνει με την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές το 2020 και αν αυτή η δημοκρατική διαδικασία συνεχιστεί τότε Πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε τη χώρα αυτή και ιδίω τα παιδιά που υποφέρουν. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, υποστηρίζω το ψήφισμα το οποίο άλλωστε έχω υπογράψει. Το 2016 κλείνουμε 25 χρόνια από την ανατροπή του δικτάτορα Μπαρέ στη Σομαλία. Ανατροπή που άνοιξε όμω, δυστυχώ ένα νέο κύκλο αίματο, ο οποίο παραμένει ανοιχτό αποτέλεσμα αυτών των 25 χρόνων της διαφυλετικής βίας είναι η Σομαλία να αποτελεί μια από τις πιο φτωχές χώρες της Αφρικής, με προσδόκιμο ζωής μόλις τα 55 χρόνια και το 1 έκτον του πληθυσμού να ζει εκτός των σύνορων της. Οι επερχόμενες εκλογές που κανονικά πρέπει να διεξαχθούν μέχρι το τέλος του έτους δεν δείχνουν να μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα. Το μείζον ζήτημα για τα κράτη της Δύσης είναι συνεπώς να κρατήσουν μακριά από την εξουσία τους Ισλάμιστέ τη Αλ Σαμπάμπ ωστόσο με τις επεμβάσεις τους οι ξένες δυνάμεις δεν επιδρούν επικοδομητικά όπως δείχνει και η εμπειρία των τελευταίων 25 χρόνων. Το καλύτερο που έχει συνεπώς να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μείνει μακριά και να μην αναμειχθεί στα πολιτικά παίγνια που δεν την αφορούν. Καμιά συμμετοχή στα βρώμικα παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα στο κέρος της Αφρικής. Αλληλεγγύη σε χριστιανούς θύματα της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Τηλιανίδης. Το μικρόφωνο σας. Ήταν πολύ παραγωγική και επικοδομητική η συζήτηση. Τη Σομαλία τη γνωρίζω. Την έχω επισκεφθεί. Έχω συναντηθεί με, τους, ε, με τον Υπουργό και άλλους αξιωματούχους. Για την εκπαίδευση ήθελα να σημειώσω πως έχω ήδη εγγράψει την εκπαίδευση σε σχέδια συνεργασίας ε, προτεραιότητας, τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε με τους εταίρους μας. Ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση για τη Σομαλία και ιδιαίτερο θα επιμένω για τα σχέδια αυτά. Η Σομαλία συχνά εμφανίζεται στα πρώτο σέλιδα σπάνια όμως με θετικό φως παρά την σημαντική βία όμως και τα προβλήματα έχουμε δει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ε, πρόοδο προς τον εκδημοκρατισμό και την εξομάλυνση θα γίνουν οι εκλογές με συμμετοχή 14.000 ατόμων που εκπροσωπούν τμήμα μόνο του πληθυσμού. Ωστόσο αυτό, όσο και αν δεν θεωρηθεί καθολική ψηφοφορία με τα δικά μας δεδομένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 135 ε, εκλεγμένοι αρχηγοί φρατριών ορίζουν τα μέλη του Κοινοβουλίου μέχρι το 2020. Η συμμετοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένως επιμείνει να Ε, διεκδικεί την δέσμευση πλευρά τη Σομαλία για συμμετοχή κατά 30% γυναικών στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο εμφύλιο ε, πόλεμο και οι συγκρούσει έχουν ε, διαλύσει αδίποτε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γυναίκε, παιδιά, άτομα με αναπηρίε έχουν συχνά πληρώσει το πιο ακριβό τίμημα των καταχρήσεων, των κακοποιήσεων της οικιακής βίας εις βάρος των γυναικών που είναι πολύ συνηθισμένα παρότι η Σομαλία έχει υπογράψει και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών πολύ συχνά τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα των ανώπλων συγκρούσεων. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν προς την υλοποίηση ενός νέου ε, συνόλου δράσεων για το 2016 που ορίζεται συγκεκριμένα, ορίζει συγκεκριμένα ως στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια με απότερο σκοπό να ενισχυθούν οι οργανώσεις των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων και η θέση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ο σεβασμός τους από τις κυβερνητικές, αστυνομικές, δικαστικές αρχές, έτσι ώστε να υπάρξει ένας χώρος δικαιοσύνης, ασφάλειας, ε, και να μειωθεί η σεξουαλική και οικογενειακή βία, να σταματήσει η ατιμορρησία των δραστών τέτοιου είδους εγκλημάτων. Για τη θανατική ποινή επίσης είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχει θέσει πέρα στο de facto moratorium η Σομαλία η ε, εκτέλεση θανατικών ποινών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπών δικαιωμάτων και της ανθρώπινας αξιοπρέπειας έχουν ε, ε, δεν δημοσιεύσει τα, ανθρώπινα, τα Ηνωμένα Έθνη σχετική έκθεση. Έχει τεράστια σημασία το θέμα αυτό προκειμένου να ε, προχωρήσουμε με την απάλληψη της ανατικής ποινής και την ενίσχυση των θερμών δικαιωμάτων στην οικοδόμηση μιας υγιούς κοινωνίας. Οι δημοσιογράφοι έχουν κέρια σημασία για μια συζήτηση σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο πέφτουν συχνά θύματα παρενοχλήσεων, προσβολών, επιθέσεων, ακόμη και συλλήψεων. Υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που ε, κλείνουν ε, με αποφάσεις κυβέρνησης και γενικά παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς καμία αίσθηση ε, λογοδοσίας. Οι θεσμοί γύρω από τη δικαιοσύνη έχουν τεράστια σημασία για την ε, υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και της δημοκρατίας στην Σομαλία. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ειρήνη για όλες τις κοινότητες της χώρας, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες έχουν υποφέρει από τις επιθέσεις Al-Shabaab. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με τη Σομαλία για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και θα συνεχίσει να το πράττει και με την νέο εκλεγήσα ηγεσία της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε.